Ε, τη λήξη της εντολής της ειδική Επιτροπής ε, για το οργανωμένο έγκλημα, τη ε, διαφθορά και την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που Εκπνέει η εντολή αυτή κανονικά στις 31 Μαρτίου του 2013 και προτείνεται παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 σύμφωνα με το άρθρο 184 του κανονισμού. Διαφωνεί κανείς? Αν όχι, Εγκρίνεται η διεύρυνση αυτή τη εντολή και η παράταση λειτουργία τη της Επιτροπής ΚΡΙΜ. Ούτως λοιπόν και αποφασίζεται. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η εντολή της Επιτροπής το 2013. Τελευταία ανακοίνωση. Ορίστε. Ο κύριος Σταφάρας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα, από ευκαιρία της παράτασης των εργασιών της ειδική Επιτροπής για κατά το οργανωμένο εγκλήματος και την νομοποίηση παράνομων εσόδων, γιατί στην οποία είμαι αντιπροεδρία, ε, αντιπρόεδρος, μια και η τράπεζα HSBC θα πληρώσει 1 δισεκατομμύρια και 200 εκατομμύρια ε, ως πρόστιμο για την ε, ε, ε προτείναμε να συσταθεί ένα κονδύλιο, ένα ταμείο, να συσταθεί ένα κοινωνικό ταμείο που θα χρηματοδοτείται από τέτοιου είδου πρόστιμα λόγω οργανωμένου εγκλήματο και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ελπίζω με την παράταση των εργασιών αυτή τη ειδική επιτροπή θα καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε τέτοιου είδου περιπτώσει. Ναι, ναι. αυτό είναι και ο στόχο, κύριε Ταβάρη, να μπορέσουν να συζητηθούν σε βάθο όλα αυτά τα οποία αναφέρατε. Τελευταία ανακοίνωση. Ορίστε η πρόεδρος της Επιτροπής. Sí, ναι, παρακαλώ, κυρία. Sí, gracias, Presidente. Sono... Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ είμαι πρόεδρος αυτή τη Επιτροπής ε, που με τη δική σας τη συνένεση ε, έλαβα ανανέωση της εντολής της. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από την Τρίτη μέχρι την Παρασκευή της προηγούμενης εβδομάδας ήμουνα στην Ουάσιγκτον και ήμουνα σε επαφή με εκπροσώπους του FBI, του Υπουργείου Οικονομικών, της Δικαιοσύνης και αυτοί λοιπόν ε, παρότι και οι ίδιοι ασχολούνται με θέματα ανακύκλωσης, ε, όλοι λοιπόν ε, αποδίδουν μεγάλη σημασία και έχουν μεγάλες προσδοκίες από την Επιτροπή μας. Εκτίμησαν ιδιαίτερα την πολύ καλή δουλειά που έχει προσφέρει η Επιτροπή μας, πάνω από 20 συνεδρίες σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη τους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αλφάνο. Λοιπόν, ευχόμαστε ε, καλή συνέχεια στις εργασίες σας. Εχθές το βράδυ ο Προεδρεύων ε, στην Ολομέλεια ε, διάβασε μια ερμηνεία του άρθρου 187 παράγραφος